Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Πρώτα έχουμε την ε, έκθεση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου. Και για όλα τα νησιά που εκεί. Η κυρία Σουίτσα έχει να πει κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτή είναι μια σημαντική έκθεση και αναφερόμαστε στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου που καλύπτει 80 εκατομμύρια ε, κατοίκους με 8 χώρες από τις οποίες ε, πέντε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άλλες είναι υποψήφιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλους αυτούς τους κανόνες. Είμαι επίσης η συγγήτρια της Επιτροπής ΕΝΒΗ και αύριο θα συζητηθεί το θέμα εκεί και θα είναι και αυτό μια σημαντική συμβολή στην έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που έχουν λάβει μέρο και έχουν βοηθήσει στην εκπόνηση αυτή τη έκθεση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την 4. 30 με 31 απορρίπτεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. «52-9 με μία αποχή γίνεται δεκτή η έκθεση. Συγχαρητήρια κυρία Σουίτσα. Και ήσασταν πολύ ικανοί στην διαμόρφωση συμβιβαστικών τροπολογιών και είχατε ένα πνεύμα πολύ θετικό και συμβαστικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 5, η έκθεση για την τωρινή πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Κυρία Λέζιν, θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στην συζήτηση αυτή, απλώς θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους σκιώδεις ε, οι συγητέ ίσως όμως θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια. Υπάρχει κάποιος κοιόδης συγητή ο οποίος θα ήθελε να πει κάτι. Κύριε Αουστρεβίτσιους, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν μια μακρά και κάπως διαδικασία. Πολλές από τις προτάσεις δεν συνείδαν με τις θέσεις μας. Υπάρχει ένας μακρός κατάλογος πληροφοριών που έχουν πολλές από αυτές αποφασιστικό χαρακτήρα. Εγώ θα ζητούσα να έχουμε μία ψηφοφορία και όχι πολλές. Θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο λογικό, λέει ο κύριος Αστρεβίτσιος. Κύριε Πρέντα. Στηρίζω και εγώ τόσο από κύριο Σαστοβίτης. Είπα ότι στηρίζω το αίτημα του Αστοβίτης. Αυτό λοιπόν που ζητάτε είναι να έχουμε μια συνολική ψηφοφορία για όλες τις τροπολογίες. Ναι, πρέπει να γίνει δεκτό φυσικά από ότι τα μέλη της Επιτροπής μας. η κυρία Λέζινγκ προηγουμένω. Και φυσικά εγώ πρέπει να αντιταχθώ σε μια τέτοια πρόταση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια τελείω αντιδημοκρατική διαδικασία. Εγώ πιστεύω πρέπει να ψηφίσουμε τι μεμονωμένε τροπολογίε. λέει η κυρία Λέζινγκ. Έχουμε λοιπόν την αίτηση από πολλές πολιτικές ομάδες να έχουμε μια κοινή ψηφοφορία. Ποιος θέλει να γίνει μια ψηφοφορία unblock των τροπολογιών υπέρ κατά αποχές είναι η πλειοψηφία. Ποιος υποστηρίζει το σύνολο των τροπολογιών που έχουν κρατηθεί, σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ, κατά αποχές Έχουν απορριφθεί λοιπόν όλε οι τροπολογίε. Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, η ηλεκτρονικά αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Η έκθεση με δύο ψήφους υπέρ και 43 ψήφους κατά και 17 αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 και ήθελα να δώσω τον, το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Πρέντα. Mr. Preda. Παρακαλώ κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Να. General budget of the European Union for the... Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2016. Πρόεδρε. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπροκ. Κοιτάξτε, σταματήστε τα πηγαδάκια αν έχετε να πείτε κάτι για τον προπολογισμό. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ. Είχα μείνει στο Αφγανιστάν. Για τον προπολογισμό θα είμαι σύντομο. Νομίζω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης εκφράζει πολύ καλά τη θέση μου. Το πήρατε χτες. Βέβαια είμαι ανοιχτό να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για τα σημεία που θεωρείτε ότι είναι σημαντικά. Για να είμαστε σύντομοι λοιπόν. Προτείνω πρώτον μια που έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης από χτες, επαναλαμβάνω θα είμαι σύντομος και προτείνω πρώτον με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να δείξουμε ότι στηρίζουμε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλουμε τις περικοπές που προβλέπονται στο σχέδιο του Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς θα προτείνω δημοσιονομικές τροπολογίες αποκατάστασης που θα χρησιμεύσουν να διατηρήσουμε τα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, προτείνω με σαφήνεια να πούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής μας Όσον αφορά λοιπόν το σχέδιο, αυτό ακριβώς θα κάνουμε τις νομικές τροπολογίες. Και όταν λέω προτεραιότητες, πρόκειται για θέματα με τα οποία συμφωνούμε νομίζω όλοι στην Επιτροπή μας. Το ένα είναι η πολιτική γυτνίαση με τι χώρε ανατολικά και νοτίω τη Ευρώπη, δεδομένου των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τη στήριξή μα. Και όχι μόνο με λόγια. Δεύτερον, η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξη της δημοκρατίας. Εδώ πρόκειται για αξίε που βρίσκονται στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Και τρίτον, θέλω με σαφήνεια να πούμε ότι δεσμευόμαστε υπέρ των υποψηφίων χωρών, διότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογο μαζί του. Και τέλο, στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, για να στηρίξουμε την Πολυστινιακή Αρχή και την Ούντρα, διότι στο σημερινό πλαίσιο χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Να λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες που προτείνω εγώ. Πέραν βέβαια από τις ε, τροπολογίες αποκατάστασης όπως σας είπα προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι εκείνη του Συμβουλίου να περάσει. Η προθεσμία για την κατασταση τροπολογιών 23 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητήλο κύριο Σπίκουλα που δέχτηκε τις προτάσεις της ομάδας μου των σοσιαλιστών όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο εισηγητής έλαβε υπόψη του κυρίως το ευάλωτο κλίμα που επικρατεί στην γειτονιά μας. Και γι' αυτό συμπεριέλαβε και τις προτεραιότητες που συμπεριλαμβάνει. Οι συνεχείς συγκρούσεις στην Μεσόγειο είναι απειλητικές και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να δεσμευτούμε περισσότερο από πλευράς μας στην ε, πολιτική γειτονία και στη Συρία και στην Ουκρανία. Χρειάζεται λοιπόν αυξανόμενη στήριξη επίσης και στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, υπέρ δηλαδή της Παλαιστινιακής Αρχής και της Ούνρα. Ως σοσιαλιστές θέλουμε να εκφράσουμε κάποιες ανησυχίες για την τελευταία παράγραφο του σχεδίου γνωμοδότησης, στο σημείο 5 δηλαδή, που λέει ότι ζητάει γραμμή προπολογισμού για τους ειδικού ε, προσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που να πάνε από το ΚΕΠΑ στην ε, εξωτερική δράση για να στηριχτεί η δράση ακριβώς της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γραμμή στον προπολογισμό για τους ειδικού εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατηρηθεί εκεί που βρίσκεται, στην ΚΕΠΑ και να μην περάσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία που χρειαζόμαστε. Επιπλέον, η ύπατη εκπρόσωπος κ. Μογερίνη ζήτησε μία μελέτη σκοπιμότητε, αλλά πιστεύουμε ότι προ το παρόν είναι καλύτερο να διατηρηθεί η σημερινή δομή και να μην αλλάξει. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο πρώτος, δίνει το λόγο. Η κυρία Λέζιν, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την έκθεσή του, μπορούμε να τον υποστηρίξουμε απόλυτα. Εμείς θα καταθέσουμε και μια τροπολογία που ζητά την αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού που αφορά την πολιτική γειτονία, όμως είμαστε λιγάκι σκεπτικιστέ λόγω του ρόλου που έχει διαδραματίσει η πολιτική γειτονία στο παρελθόν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση του κοινωνικού πλαισίου και του πλαισίου υγειονομικής περίθαλψης και όχι μονάχα του επιχειρηματικού κλίματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι όλα αυτά που γίνονται στην άμεση γειτονιά μας, είτε προς τα ανατολικά είτε προς τα νότια, πρέπει να είναι μια σαφής προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό του 2016. Και η ομάδα του, της Άλντε υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση ότι πρέπει να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι για να ενισχυθούν οι θετικές εξελίξεις στην άμεση γειτονιά μας και να τύχουν σε αυτοί οι πόροι και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας τους θα πρέπει να έχουν μια προεξάχουσα θέση στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, όπως είπα και στην αρχή, η ημερομηνία προθεσμία για την υποβολή τροπολιών 23η Ιουλίου. Υπάρχει και συνάντηση με τον κύριο Φερνάντες βέβαια, σε λίγες ώρες προκειμένου να συζητήσουμε. Οπότε σας δίνω ραντεβού μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για την 31η Αυγούστου προβλέπεται η ψηφοφορία. Σωστά πρόεδρε? Υπάρχει αντίθετη απόψη για την ε, στιγμή της ψηφοφορίας, εάν όχι. Έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα αγαπητοί συνάδελφοι. Η αντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα έρθει στις 11. Μπορούμε να συζητήσουμε το Ιράν. Δεν βλέπω τώρα αν υπάρχει ε, μεγάλη παρουσία, αλλά θα έρθει και η κυρία Μογκερίνη να κάνουμε μια συζήτηση μαζί της. Αυτό προβλέπετε. Ή θέλετε να κάνουμε τώρα μια συζήτηση ή μπορούμε να κάνουμε μια διακοπή για καφέ. Μια διακοπή καφέ, αλλά σας παρακαλώ, επειδή θα έρθουν συνάδελφοι από την Ουκρανία, να επανέλθετε στις 11 και να φέρετε και μερικούς συναδελφούς από τις πολιτικές σας ομάδες. Θα είναι κρίμα, θα είναι λυπηρό να είναι άδεια τα έδρανα της Επιτροπής μας όταν έρχονται οι άνθρωποι από την ε, Ουκρανία. Έχουν πάρα πολλοί φύγει για διακοπές και στο μέλλον θα ζητήσω να μην υπάρχει τέτοια κοινοβουλευτική εβδομάδα μετά από την Ολομέλεια. Στο παρελθόν είχα μια έκθεση στη Συνταγματική Επιτροπή και ήμουν ο μόνος ο οποίος ήμουν παρόν από την πολιτική μου ομάδα και αυτό συμβαίνει σε πολλές επιτροπές αυτή τη εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι η τελευταία εβδομάδα, η εβδομάδα Ολομέλειας του Ιουλίου, να υπάρχει ίσως μια εβδομάδα επιτροπών πριν από την Ολομέλεια, αλλά όχι μετά από την Ολομέλεια. Αλλά αυτή η εβδομάδα πάντως είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τι γίνεται. Ε, πολλές φορές έχουμε και τις οικογένειες μας να σκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στις Ευχαριστώ. <laughs> Υπότιτλοι AUTHORWAVE στο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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 AUTHORWAVE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 Υπότιτλοι Authorwave Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Wir sollten anfangen. Ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς που είναι εδώ παρόντες. Καλώς ορίζουμε εδώ τα μέλη μιας μεγάλης αντιπροσωπείας από την Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν πολλούς αναπληρωτές υπουργούς που είναι εδώ παρόντες. Η κυρία Γνιούντιοκ είναι η, η επικεφαλής αντιπροσωπείας που είναι υπουργός ε, επικρατείας του επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού και επίσης έχουμε την ε, αρμόδια για τα ευρωπαϊκά θέματα και θα μας κάνει μια παρουσίαση στη συζήτηση και θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στην κυρία Κάλλας, η οποία πρέπει να φύγει βέβαια σύντομα. Στις 11.30 θα πρέπει να φύγει, ώστε θα της δώσουμε και αυτή την ευκαιρία να μπορέσει να λάβει το λόγο ως ε, αναπληρωτής πρόεδρος της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας. Σας παρακαλώ λοιπόν κυρία Υπουργέ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα και εκ μέρους της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας να έρθουμε εδώ σήμερα και να συναντηθούμε μαζί σας. Είναι δύσκολη καιρή για την Ουκρανία και συγχρόνως προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, αλλά συγχρόνως να προχωρήσουμε σε βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και μεταρρυθμίσεις στη δημόσια ζωή. Γνωρίζετε ότι για μας είναι πολύ σημαντικό ότι αρχίσαμε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής για τη Σύνδεση, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εφαρμόσουμε και να συντονίσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη αυτή. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο υπογράψαμε πριν από ένα χρόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμφωνία αυτή Σύνδεσης. Η διαδικασία τώρα συνολικών και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης και είμαστε αφοσιωμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως εκείνους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ουσιαστική στήριξη που έχουν δώσει μέχρι τώρα στην Ουκρανία και αυτό φάνηκε και πριν από 1,5 χρόνο από τα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντάν. Γνωρίζετε ότι αυτή τη βδομάδα, χτες συγκεκριμένα, αρχίσαμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης. Είναι ένα εργαλείο που θέλουμε να δουλέψει. Και πέρυσι βέβαια το Δεκέμβριο είχαμε το Συμβούλιο Σύνδεσης και είχαμε και συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αρχίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να θέτουμε σε εφαρμογή τις υποχρώσεις μας από τη Συμφωνία αυτή σύνδεσης. Θέλω να επιβεβαιώσουμε την ε, δέσμευσή μας αλλά και την αμοιβαία δέσμευση που υπάρχει μεταξύ μας όσον αφορά την εφαρμογή των, ε, προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας. Όσον αφορά την επικύρωση και τη διαδικασία επικύρωσης τώρα από όλες τις χώρες μέλη της συμφωνίας αυτής της σύνδεσης, την παρακολουθούμε και προσβλέπουμε σε πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης. Εμείς περιμένουμε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2016 θα μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε πλήρως. Όλοι οι πολίτες στην Ουκρανία αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνία αυτή, σε αυτά τα πλαίσια, αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο που μας έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ε, Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά από πλευράς των Ουκρανών παραγωγών. από 1η Ιανουαρίου 2016, όπως σας είπα, θα τεθεί πλήρως εφαρμογή και προσβλέπουμε στη δικιά σας στήριξη για το πρόγραμμα δράσης μας όσον αφορά την ελευθέρωση. Η Ουκρανική κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε πιο εντατικές εργασίες για να προχωρήσει και έκθεση όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό ελευθέρωσης των συναλλαγών. Ελπίζουμε αυτό το μέσο να το έχουμε στη διάθεσή μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το εργαλείο αυτό θα αποτελέσει και το κύριο αποτέλεσμα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση που θα δείχνει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταρρυθμίσεις μας και θα ανοίγει την πόρτα στους Ουκρανούς πολίτες. Είμαστε επίσης ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της που μας έδωσε την ευκαιρία να υπογράψουμε και τη συμφωνία για την αεροπλοΐα. Έχουμε έτσι πρακτικές επιτυχίες όσον αφορά τις διμερείς μας σχέσεις. Τη συμφωνία αυτή τη στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ως δικιά μας επιλογή μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Κρυμαία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά την Ευρωπαϊκή Ομάδα που στήριξε επίσημα την Ουκρανία σε όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως χώρα. Ελπίζω ότι η άτυπη αυτή ομάδα θα γίνει επίσημη και θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική και να εκπροσωπεί και όλα τα εθνικά κοινοβούλια από όλες τις χώρες μέλη. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης και καλωσορίζουμε το νέο σχέδιο που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από κοινού θα το εφαρμόσει με την Ουκρανία και που έχει να κάνει με την αμοιβαία συνεργασία. Ως κυβέρνηση έχουμε δεσμευτεί υπέρ αμοιβαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Χαίρομαι πολύ που σήμερα δεν βρίσκομαι μόνη μου στο Κοινοβούλιο. Έχω μια κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνη για την για τη σχέση μας με την Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι άνθρωποι υπεύθυνοι για τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις, για τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτές είναι δύο κατευθύνσεις που πρέπει να προχωρήσουν, να ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές μας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε εμένα προσωπικά αλλά και σε ολόκληρη την ομάδα, τους συνεργάτες μου δηλαδή και εμένα που με υποδεχτήκατε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Ως αντιπρόεδρος της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να είμαι εδώ ενώπιον σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ουκρανίας θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις. Η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντική για την αμοιβαία μας συνεργασία για να μπορούμε να καταλάβουμε η μεν και η δε τις ανάγκες της άλλης πλευράς και μόνο με την συνεργασία μας θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης μπορεί να προχωρήσει με ομαλό τρόπο. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες πρόσφατα ότι κάποιες από τις, κάποιες από τις πρόοδους που είχαν επιτευχθεί μπορούν να αναστραφούν. Μιλώ για νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο που θέλουν να αναστρέψουν και να ακυρώσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις Κατανοώ όμως ότι η θέση του, της κυβέρνησης όπως και της Βουλής είναι δύσκολη. Πρόσφατα στις αρχές Ιουλίου, ενώπιον της Βερχόβνα Ράντα του Κοινοβουλίου, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, παρακολουθήσαμε και τη διαδικασία των συζητήσεων που έλαβαν ε, χώρα για μερικά από τα δύσκολα νομοθετήματα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορεί να είναι πραγματικά οδυνηρές στο άμεσο μέλλον είναι δύσκολο να τις εξηγήσουμε στο λαό της Ουκρανίας. Πρέπει όμως να δούμε τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα. Είναι κέρδιες αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει η Ουκρανία να επανέλθει στην ανάπτυξη και να γίνει μια ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία θα πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν με αποτελεσματικό τρόπο και θα απαρμοστούν πλήρως και η κοινή γνώμη καταλαβαίνει ε, την ανάγκη αυτών των μεταρρυθμίσεων για ένα θετικό αποτέλεσμα εν καιρό και από τη δική μας πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό η, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια θετική συμβολή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν περάσει αντίστοιχες διαδικασίες μεταρρύθμισης από τις οποίες μπορούμε να εμπνευστούμε κι εμείς. Αυτή η συνεργασία λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, εμπειρία που έχουμε στην Ουκρανία προς το καλό όλων. Προσβλέπω λοιπόν στην συζήτηση μαζί σας και στη συνεργασία μαζί μας. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much and uh, very warm welcome to you all. ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε όλοι και πρώτα πρώτα να σας διαβιώσουμε για κάτι ότι όχι μόνο από πλευρά του ΕΛΚ αλλά οι περισσότερες πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται εδώ συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την προσέγγιση, την γενικευμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία αλλά επίσης και για το πώς αντιδρούμε στην ρωσική κριτικότητα και θέλουμε την παράταση ε, των κυρώσεων όπως έγινε αυτό τον Ιανουάριο και αυτό αποδεικνύει την άποψή μας. Γι' αυτό λοιπόν και είναι σημαντικό σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνουμε συσπηρωμένοι και να αντιτιθέμεθα ε, σε αυτήν την ρωσική επίθεση. Τώρα όσον αφορά το θεματολόγιο σε σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης και όλες αυτές τις προσπάθειες που έχετε αναλάβει. Εγώ, αναφαντών, σας υποστηρίζω και με αυτό να έχει γίνει πιο νωρίς να φτάσετε σε ένα σημείο τόσο ώστε να έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για την κατάργηση της θεώρησης διαβατηρίου για τους ε, πολίτες της χώρας. Είναι συναισθηματικό το θέμα, πολιτικό, αλλά και από τεχνική ακόμα πλευρά. Έτσι μπορούμε να αποδείξουμε τον δεύτερο τρόπο αυτή την υποστήριξή μα και αυτό να, μπορεί να το νιώσει ο, κάθε Ουκρανό πολίτη. Επίση, κάτι θέλω να ρωτήσω όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη δέσμευση. Ε, πριν από τέσσερις μήνες προείδρευα σε εκείνη την ε, αποστολή αρρωγή στο Κίεβο και θέλαμε να καλύψουμε κάποιες, ε, κάποιους τομείς ιδίως όσον αφορά το, το, το, το δίκαιο που διέπει τη δράση του Γενικού Εισαγγελέα, κάποια άλλα θέματα ιστορικής ασφάλειας. Για αυτούς τους τέσσερις τελευταίους μήνες, τι έγινε, μπορεί να μας εξηγήσετε πώς η κατάσταση των πραγμάτων, τι μέτρα έχετε θεσπίσει, ε, Πώς, πώς, αξιολογείτε τη δική μας συμβολή, τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε περαιτέρω. Τι λέτε για αυτή την ε, αποστολή αρρωγής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Παντζέρη. Και εγώ να ευχηθώ καλώς όρισαν οι προσκεκλημένοι μας. Δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε το ότι δεσμευόμαστε για πλήρη συνεργασία όσον αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης. Κυρίως όσον αφορά εκείνα τα κεφάλαια που θεωρούμε ότι είναι τα πιο σημαντικά εκείνα που αφορούν την ε, ε Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και όσον αφορά τους δασμούς επίσης αλλά και την κινητικότητα των εργαζομένων όπως και τα της θεώρησης διαβατηρίων. Επομένω, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι μα ενδιαφέρει το να υπάρξει πλήρη συνεργασία και θέλουμε να υποστηρίξουμε τη χώρα. Επίση, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι θα πρέπει η Συμφωνία Σύνδεση να υλοποιηθεί και όσον αφορά το πολιτικό τμήμα τη, αλλά κυρίω όσον αφορά τα συγκεκριμένα κεφάλαια αυτή. Και έτσι, αυτό θα γίνει δυνατό όταν έχουμε την διαδικασία της μεταρρύθμισης θα πρέπει να γίνουν αυτές οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις ακριβώς όπως είπε η κυρία Κάλλας. Βεβαίω θα είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει τον πληθυσμό αλλά είναι αναγκαίο. Και έτσι να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εφαρμογής της συμφωνίας. Τώρα, πέστε μου σας παρακαλώ, τι πρεσβεύετε πάνω σε αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην ε, ολοκλήρωση και εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Έχουμε τώρα το θέμα του τι θα γίνει με την Ρωσία και την Κρυμαία. Νομίζω ότι και σε εκείνο το μέτωπο θα βοηθήσει η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων, οπότε γι' αυτό και εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να συνεργαστούμε 100%. Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε έντονα ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρώσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ βρίσκομαι. Είμαι από την τρίτη σε μέγεθος πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πολύ φίλοι της χώρας σας, της Ουκρανίας. Εγώ προσωπικά παρατηρώ από το 2002 το τι γίνεται στην Ουκρανία, όταν κάποιος δημοσιογράφος με ρώτησε τη Wall Street κατά πόσο έχει ευρωπαϊκή προοπτική χώρα. Ε, είναι εδώ ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Βόλσκι και εγώ είμαστε παρόντες στην ε, Πορτοκαλία Επανάσταση και έχουμε συμμετάσχει στην Ουκρανική διπλωματία. Ο κύριος Πούτιν έκανε λάθος υπολογισμούς προσαρτίζοντας τμήμα της επικράτειάς σας. Και τώρα έχει καταλάβει 5% της επικράτειάς σας και ξοδεύει πάρα πολλούς οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους για να διατηρήσει αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες δεδομένης και της τόσης της τιμής του πετρελαίου. Η κυβέρνηση δικιά σας από την άλλη πλευρά πρέπει και εκείνη να εξοπλίζεται για να προστατεύσει την επικράτειά σας. Εμείς στηρίζουμε όλες τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην προσπάθεια του Πούτιν να δημιουργήσει το διάδρομο αυτόν και να μεγαλώσει και να κάνει πιο ευνοϊκή την κατάσταση προς αυτόν, την καταδικάζουμε και συμμετέχουμε και εμείς στις διπλωματικές προσπάθειες για να μην πετύχει. Και είμαστε υπέρ παρετέρω κυρώσεων. Χτες έμαθα ότι παρά τον πόλεμο που λαμβάνει η χώρα στα ανατολικά της χώρας σας, εσείς ετοιμάζεστε να στείλετε ε, στο Αφγανιστάν κάποιους δικούς σας στρατιωτικούς για να εκπαιδεύσουν εκεί τον κόσμο. Πολύ θαραλέω εκ μέρους σας θα έλεγα αυτό. Σλάβα Ουκραίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ. Ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατα μονάχα εγκρίναμε την έκθεση για την ε, Μαύρη Θάλασσα και αναφέραμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας. Είναι κάτι που πρέπει και εσείς να αντιμετωπίσετε τους επόμενους μήνες. Για μας η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι κομμάτι της δικής μας ασφάλειας, ασφάλειας της κεντροανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα επίσης να μας εξηγήσετε τι θέλετε εσείς. Να μας εξηγήσετε τις ανάγκες σας. Η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται σε αλληλεγγύη. Θα έχετε ακούσει για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα πρέπει να εγκρίνει η Ουκρανία αυτό το κεκτημένο στα πλαίσια της προσέγγισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μας πείτε όμως και τι περιμένετε. Είσαστε η έκτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη, μια μεγαλύτερη χώρα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι χώρες πρέπει να εκφράσουν τις προσδοκίες τους. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, χάσαμε μια ευκαιρία όταν ζήτησε ο πρόεδρος Ποροσέγκο να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο συγκεκριμένες αιτήσει για το τι μπορεί να γίνει από τη διεθνή κοινότητα για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ουκρανία. Η Ανατολική Ουκρανία είναι εκεί που αποφασίζεται το μέλλον της ειρήνης για την Ευρώπη. Έχω να κάνω και ένα ακόμα σχόλιο. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι κέριος. Δεν θα υπάρξει μέλλον για τη δημοκρατία αν μπορεί κανείς να αγοράζει τους δημόσιους λειτουργούς. Εάν η κοινή γνώμη δεν είναι πεπισμένη ότι υπάρχει κράτος δικαίου, αν οι αποφάσεις της κυβέρνησης δεν υπαγορεύονται από τις ανάγκες του κόσμου, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μια άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η εμπειρία των άλλων χωρών στην κεντροανατολική Ευρώπη. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να είναι πεπισμένος ο λαός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι προς το συμφέρον τους. Δεν πρέπει να είναι μια εφαρμογή μιας αφηρημένης ιδεολογίας, πρέπει να είναι πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Πράγματι είναι δύσκολες κινήσεις, δεν είναι εύκολο να βγει κανείς από την κομμουνιστική νοοτροπία, το ξέρουμε από τη δική μας ε, εμπειρία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να σας βοηθήσουμε και ενθαρρύνοντάς σας πάντα να δράσετε προς το καλύτερο συμφέρον της χώρας σας και περιμένουμε να μας αναφέρετε τι περιμένετε από εμά γιατί η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. κύριο Ευχαριστώ λοιπόν του εκπροσώπους της Ουκρανίας που έρχονται στι Βρυξέλλες. Είναι ιδιαίτερα καλόδεκτοι και δεν είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε σε επαφή, αλλά κάθε φορά είναι μια μεγάλη χαρά για μα γιατί μπορούμε να έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Χαιρετίζω το γεγονό ότι η αντιπροσωπεία τη Ουκρανία απαρτίζεται από νέου ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια νέα γενιά να αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέλλον της χώρας της. Αυτό είναι και για μας ένα πολύ καλό μήνυμα οι άνθρωποι αυτοί είναι αποφασισμένοι να υπηρετήσουν τη χώρα τους μέσα από την πολιτική και τη δημόσια διοίκηση. <clears throat> Είναι πάρα πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ουκρανία. Και αυτό είναι το τίμημα δύο δεκαετιών που δεν έγιναν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει έφορο το έδαφος για μεταρρυθμίσεις και μετά να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Η Ουκρανία έχει πάρα πολλούς περιορισμούς γιατί βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Πάνω από 20% των εθνικών πόρων θα πρέπει να αφιερωθούν στο, στη διεξαγωγή του πολέμου λόγω της εισφολής της Ρωσίας στην Κρυμαία και την νοτιοανατολική Ουκρανία. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να γίνουν όλα αυτά. Συγχρόνως να κάνετε μεταρρυθμίσεις. Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι είστε ένα καλό παράδειγμα ακόμα και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν είναι έτοιμα να κάνουν κινήσεις και να πάνε τις απαραίτητες αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις και να τις εφαρμόσουμε. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα και πιστεύω ότι η Ρωσία δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Η Ρωσία χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι μια απειλή για τον εαυτό της. <laughs> Όσο λοιπόν προχωράτε θετικά δείχνετε και το σωστό δρόμο στην Ρωσία. Και για σένα Νατάλια και την ομάδα σου θέλω να πω τα εξή. Από την πρόσφατη ε, συνέντευξη τύπου του, πρόεδρου, του Πρωθυπουργού Γιατσενιούχ πρωτού πάει στις ΗΠΑ είπε ότι εμείς ως κυβέρνηση έχουμε στείλει στο Κοινοβούλιο στην Βεχόβνα Ράντα, στο Κοινοβούλιο πολλές ε, νομοθετικές προτάσεις, οι οποία όμως καθυστερεί κάπως για την έγκριση αυτής της νομοθεσίας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τη συνεργασία μεταξύ του εκτελεστικού τομέα και της νομοθετικής εξουσίας και σε ποιο βαθμό είναι σωστά ενορχιστρωμένη αυτή η διαδικασία για την έγκριση της νομοθεσίας. Και επειδή είσαστε στις Βρυξέλλες, είναι γεγονός ότι έχετε κινητοποιήσει πάρα πολλούς πόρους και έχουμε την ε, εκπρόσωπο της ομάδος ε, συνεργασίας και αυτό είναι ιδιαίτερα καλόθεκτο. Πώς όμως εκτιμάτε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την αρρωγή και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους, δηλαδή μια ευρωπαϊκή μεταρρυθμισμένη και καλά ενσωματωμένη Ουκρανία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουνα πρόσφατα στο Κίεβο και θέλω να πω το εξή. Εγώ είδα να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Είναι διαφορετικό το πνεύμα των πολιτικών με τους οποίους μίλησα. έχουν αναλάβει μεγάλες ευθύνες και έχουν αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο πλέον το πολιτικό στερέωμα. Είναι δεσμευμένοι για περισσότερες μεταρρυθμίσεις και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης έχει αποτελέσει μια μεγάλη πρόοδο. Δεν μιλάμε μονάχα σε επίπεδο πολιτικών αυροφροσινών και ασαφών ε, στόχων έχουμε συγκεκριμενοποιήσει την συνεργασία μας επί τη βάση κοινών αρχών και αξιών. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια καλύτερη απόφαση για να κινηθεί η Ουκρανία προς μια πολιτική η οποία θα είναι σταθερή συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης για το γεγονός ότι με την κοινοβουλευτική συνεργασία έχουμε πια ένα πιο θεσμοποιημένο και σταθερό πλαίσιο. Και εμείς θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όμως παραμένουν ακόμα εκρεμή. Και ε, αυτά πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενο συζήτησης όταν υπάρχουν διαφορέ. Υπάρχουν τομεί όπου υπάρχει δυνατότητα προόδου και θέλω να το επαναλάβω. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η ευκυβερνησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία πολιτικά και σε επίπεδο ουσίας για να μπορέσει όμως να υπάρξει αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη μια ευκυβερνησία όχι μονάχα στην Ουκρανία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει καλή διακυβέρνηση στην Ουκρανία και να χρησιμοποιήσει καλά τους εθνικούς της πόρους η Ουκρανία. Να προχωρήσει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υπάρξει πραγματική ποιοτική αναβάθμιση της πολιτικής στην Ουκρανία Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας. Και επίσης πρέπει να υπάρξουν και οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε σχέση με το εξωτερικό της Ουκρανίας. Χαίρομαι λοιπόν για την μελλοντική μας συνεργασία και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Η Λίδια... Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω να καλωσορίσω εδώ τους φιλοξενουμένους μας. Όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική προοπτική της Ουκρανίας, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση πολιτική, οικονομική που είναι δύσκολη. Έχουμε ακούσει επίσης ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τις διοικητικές αλλαγές μέσω του, της Βουλής της Ουκρανίας. Όμως όλα αυτά οδηγούν σε ταραχές στην κοινωνία. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ή υπάρχει ελπίδα. Ε, για σας που έγκυται η ελπίδα για την Ουκρανία. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα πάνε πιο εύκολα ή θα βρεθούμε σε διέξοδο στην Ουκρανία. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλό να συνδυτοποιεί ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Γιατί αν πρέπει να δράσουμε, τότε πρέπει να δράσουμε έγκαιρα και όχι να αντιδράσουμε μόνο κατόπιν εορτής. Πρέπει δηλαδή να προλάβουμε μια κρίση προτού αυτή λάβει χώρα. Αυτό ακριβώς σημαίνει στο κάτω-κάτω και εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλωσορίζω τους συναδέρφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η έκτακτη κατάσταση στην Ουκρανία συνεχίζεται εξαιτίας του πολέμου στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Συγχρόνως όμως, και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να στηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία για να επικαιρώσουμε πλήρως τις συμφωνία σύνδεσης, όλες οι χώρε μέλη δηλαδή. Για μένα προσωπικά είναι μια απογοήτευση το ότι δεν έχουν ακόμα επικυρώσει όλες οι χώρε την ε, συμφωνία αυτή πριν τη διάσκεψη της Ρήγα. Δεύτερον, τα θέματα ελευθερίας. Πιστεύω ότι θα λυθούν οι κατάλληλες αποφάσεις πριν τα τέλη της χρονιάς. Δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα της ε, μη αναγκαιότητας θεωρήσεων. Πιστεύω ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ισχύσει το καθεστώς αυτός, αυτό, να μην χρειάζονται δηλαδή θεωρήσεις, βίζα, οι πολίτες της Ουκρανίας για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει σχέδιο στην Ουκρανική κυβέρνηση για μαζικές ιδιωτικοποίησεις, πάντως είναι σημαντικό εμείς να ενθαρρύνουμε ευρωπαϊκές εταιρείες να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ιδιωτικοποίησεων. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για το οικονομικό, τα χρήματα, τις επενδύσεις, πρόκειται και για το know-how. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει και μια νοτροπία εργασίας. Αν κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στην Ουκρανία, τότε πρέπει να υπάρξει μια νέα νοοτροπία στις ε, επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αυτή τη διαφορά. Οπότε ενθαρρύνω και τις δύο πλευρές και την Ουκρανική να είναι όσο γίνεται περισσότερο ανοιχτή προκειμένου ε, επιχειρήσεις να επενδύσουν και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησεων και ενθαρρύνω τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς. Όσον αφορά τώρα την οικονομική στήριξη και αρρωγή. Κοίταξε, στη διάσκεψη για την πολιτική γειτονία 1,8 δις ευρώ αποφασίστηκαν να δοθούν ως ε, στήριξη στην Ουκρανία. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάπου 25 με 30 δις χρειαζόντουσαν, αλλά αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στις μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς και άλλων, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Η Ουκρανία βέβαια είναι αυτή η οποία θα εφαρμόσει τα μέτρα. Όλοι ξέρουμε ότι και για την εισαγγελία υπάρχουν ακόμα δυναμίες και ε, σε επίπεδο δικαστικού σώματος γενικότερα. Οπότε πρέπει να πετύχουμε όλοι μαζί. Και θα ήθελα και εγώ να δω την Ουκρανία μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το πετύχουμε. Συγχρόνως όμως, ξαναλέω, ότι πρέπει πάνω απ' όλα να σταματήσουμε τον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει εδώ πέρα μια παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Ευχαριστώ. Σαρισβόλσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, uh time... Πρόεδρε. Για να δούμε πώς μπορεί κανεί να ολοκληρώσει. Τι μπορεί να μπορεί κανεί να προσθέσει σε όλα αυτά τη θερμή υποδοχή, τη, τη, την, το γιατί βέβαια θα πρέπει να μιλήσουμε και για κάποια συγκεκριμένα πράγματα την άλλη μεριά, όπως ας πούμε το, το κοινοτικό κεκτημένο, την ε, ε, μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο των κανόνων για το, σχέδιο ε, της ε, σύνδεσης, οπότε θα πρέπει και εσείς να προχωρήσετε και να έχουμε αυτές τις εκθέσεις πρόοδου που θα επισέλθουν στις λεπτομέρειες. Επομένω τώρα ήρθε η ώρα για έργα, για συγκεκριμένα πράγματα και όχι πια για γενικολογίε. Τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για τη χώρα. Αυτό διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση. Και στο Συμβούλιο και στα δεσμικά όργανα, αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση, καμία αντίδραση από την κυβέρνηση της χώρας. Εκεί υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το πώς θα υπάρχει συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα πρώτα με το νέο Υπουργείο, νέα υπηρεσία ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ε, η υπηρεσία της αρρωγής και πώς θα είχαμε για τη διαδικασία της σύνδεσης αποτελέσματα. Νομίζω ότι η συνδεδεμένη χώρα, όπως η δική σας, θα έπρεπε να τοποθετηθεί, να αντιδράσει σε αυτά που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε και σας ερωτώ, τι γίνεται με τον συντονισμό, τι γίνεται με τον συντονισμό με τις δομές της ε, βοήθειας προς την ε, χώρα, πέραν των ε, ατομικών συνεργασιών με κάποιους υπουργούς και τελικά υψηλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης. Τώρα κάτι άλλο. δεν είναι σαφές το πόσο και αν συνεργάζονται οι υπηρεσίες της ε, κυβέρνησης με τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Επίσης, ποια είναι η σχέση μεταξύ του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, γιατί είχαμε και κάποιες μεταβολές. Και των ε, δομών του δικού σας φορέα. Επίσης, τι γίνεται για τις σχέσεις με άλλες συνδεδεμένες χώρες. Για άλλες συνδεδεμένες χώρες. Τι λένε για αυτή την ε, διαδικασία ε, παρακολούθησης που οργανώνει η Επιτροπή μας. Θα πρέπει να συναντώμεθα συχνότερα και όχι θα είμαι εισηγητής. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πέραν των ε, ευγενιών, των ε, γενικολογιών, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε στη δουλειά μας και θα πρέπει να επισέλθουμε σε κάποια θέματα πιο ομά, πιο συγκεκριμένα, πιο ενδελεχώς να δούμε τι γίνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που θα πρέπει να ενταχθούν στο ε, ιστορικό σας δίκαιο, να δούμε τι θα γίνει με την διάθεση των χώρων, να δούμε ποιες είναι οι άρεστες πρακτικές και επίσης, πέστε μα, εάν έχετε κάποιο παράπονο από το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι θεμητό σαν παράπονο, Μπορεί να είστε πάρα πολύ ευγενεί να μην το αποφεύγετε, να το πείτε, αλλά πρέπει να το πείτε που υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο ε, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να ε, συζητούμε μαζί σας τα θέματα και το τι καταφέρνετε εσείς με την Συμφωνία σύνδεση, αλλά και το τι, κάνει, ε, τι κάνουν οι υπηρεσίες οι δικές μας. Γι' αυτό και υπάρχει η ειδική task force, η ειδική γενική, η γενική διεύθυνση που ασχολείται με αυτό γιατί πολλές φορές ε, τα θεσμικά όργανα είναι μακριά από την πραγματικότητα. Οπότε η δική μας δουλειά είναι να παρακολουθούμε και εσάς και εκείνους. Οπότε να μην διστάσετε και να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια τι γίνεται. Γιατί μπορούμε κάλλιστα να τα πούμε και κλεισμένα των θυρών χωρίς κοινό και χωρίς την παρουσία της Κομισιόν. Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για αποτυχία. Θα πρέπει να πετύχει συμφωνία σύνδεσης και θα πρέπει να τα καταφέρουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε διακεκριμένοι Ουκρανοί φίλοι, καλώ ήρθατε και θα σταματήσω εδώ. Δύο ερωτήσει. Πρώτον, πώς εκτιμάτε ότι προχωράει η εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ, γνωρίζοντας ότι για ορισμένα όπλα όπως είναι, για ορισμένα μάλλον στοιχεία εξοπλισμού όπως τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, η αποστολή αυτή δεν έχει την ικανότητα παρακολούθηση. Πώ θα πετύχουμε του κοινού στόχους μας και δεύτερον, τι προτείνεται να κάνει η Ευρώπη για την Κρυμαία, γνωρίζοντα ότι η Κρυμαία δεν περιλαμβάνεται σε καμία συμφωνία, ούτε την πρώτη του τη δεύτερη του Μίνσκ και βάσει του διεθνούς δικαίου η Ουκρανία, η Κρυμαία μάλλον, είναι τμήμα της Ουκρανίας και πρέπει να τα επαναλαμβάνει η Ευρώπη σε κάθε ευκαιρία. Τέλος, θέλω να πω ότι ως Ρουμάνος και Σοσιαλιστής πρέπει να υπογραμμίσω την πλήρη υποστήριξή μας στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και στο λαό της Ουκρανίας που προχωρούν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις κάτω από πολεμικές συνθήκες, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και πάντα πρέπει να τονίσουμε την αναγνώρισή μας για αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Yeah. Uh, I Ένα ερώτημα μονάχα. Θα μπορέσει η κυβέρνησή σας να αποφοπλίσει τον δεξιό τομέα. Ε, thanks very much. Ε, ε, very... Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Θα είμαι σύντομο. Όντω έχετε δίκιο ότι είναι χωρί προηγούμενο αυτή η πρόκληση και έχουμε βέβαια αυτή τη ρωσική πίεση που λαμβάνει πολλέ μορφέ και έχουμε και τι εσωτερικέ προκλήσει για την μεταρρύθμιση. Οπότε εκτό του ότι είναι χωρί προηγούμενο αυτή η πρόκληση και εμεί αντίστοιχα σα έχουμε προσφέρει βοήθεια χωρί προηγούμενο ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ω Κομισιόν. Επίση Αναφέρατε την μακροοικονομική βοήθεια, αυτά τα 1,8 δις ευρώ. Και ακριβώς εμείς μέσω του Διεθνούς του Ταμείου ε, ε, συμμετέχουμε σε αυτά τα 17,5 δις αρρωγής. Οπότε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σας δίνουμε υπομορφή ε, δανείων και δωρεών. Ε, σαν δημοσιονομική αρρωγή, σαν τεχνική αρρωγή. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία όσον αφορά τις συνεργικές προμήθειες. Οπότε ε, έτσι, τουλάχιστον φέτος το χειμώνα, έχετε εξασφαλίσει ενέργεια. Επίσης, συμμετέχουμε στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για εμπορικά ζητήματα μεταξύ ημών και της Ρωσίας. Και επίσης, σε, διάφορες, ε, σε διάφορα άλλα επίπεδα, όπως επίσης και ότι γενικότερα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη χώρα. Έχει δίκιο ο κύριος Αρεσβόλσκι. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά το κοινωνικό κεκτημένο. Όμως, αυτό δεν είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι ε, κάποιε άλλε ανταλλαγέ, συστημικέ αλλαγέ μάλλον συστημικέ, όπω η μεταρρύθμιση τη ε, διοικητική μηχανή, τη ε, δικαιοσύνη και η καταπολέμηση τη διαφθορά, γιατί αν δεν λειτουργούν όλοι αυτοί οι τομεί, δεν γίνεται τίποτα. Δεν, δεν είναι δυνατόν να, αν δεν υπάρχει κράτο δικαίου, τότε όλα τα πλούτη του κόσμου δεν θα σα φτάσουν, γιατί έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Εκτό από τα τεχνικά ζητήματα θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και στους τομείς που προαναφέραμε και εκεί θα δούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Οπότε μπορούμε να παράσχουμε σύμβουλες, να παράσχουμε εμπειρογνωμοσύνη αλλά και τη δημοσιονομική βοήθεια. Πάντως και εσείς θα πρέπει να επιδείξετε πολιτική βούληξη και επίσης προθυμία να υλοποιήσετε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις. Μπράβο που θεσπίσατε την κατάλληλη νομοθεσία για πολλούς τομείς. Αυτό είναι ένα σωστό θεμέλιο. Αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί η υλοποίηση αυτών των νομοθετημάτων και θα πρέπει ίσως να συγκροτήσετε κάποια θεσμικά όργανα και θα πρέπει επίσης να έχετε την κατάλληλη εκτελεστική νομοθεσία. I'll try to answer Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα συνδυάζω γιατί κάποια από αυτά επικαλύπτονται. Αν μου επιτρέπετε ξεκινώ με την απάντηση στον πολωνοφίλο μου τον Σάριο Βόλσκι. Ξέρω ότι έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στη χώρα μας και έχει πάντα αντιδράσει σε όλες τις ε, προσπάθειες που έχουμε κάνει στην κυβέρνησή μας. Συνεχίζει τα πολωνικά. Μερικές φορές λοιπόν είναι μια πρόκληση και αυτά που λέτε, αλλά είναι πάντα σωστά αυτά που λέτε και μας βοηθούν να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις μας. Συγγνώμη λοιπόν για την παρέκφαση στα πολωνικά. Θα μιλήσω για την τεχνική αρρωγή, γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές το ερώτημα του πώς η Ουκρανική κυβέρνηση εκτιμά και αξιολογεί τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ελέγχθη από τον κύριο Μπάους. Η Ουκρανία έχει δύο κυρίως αιτήσει σε μακροοικονομική χρηματοδότηση που έχουν κατατεθεί και έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο για την τεχνική αρρωγή πρόκειται για χορηγήσεις προς την ε, Ουκρανική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν σε στόχο να βοηθήσουν μέσα προτε... κατά προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις. Εφέτος είχαμε 5 ή 6 προγράμματα για την υποστήριξη του κεντρικού προπολογισμού με ένα ειδικό εργαλείο για να προωθηθεί μεταρρύθμιση σε τομείς όπως είναι οι υποδομές, η δημόσια διοίκηση ή μεταρρυθμίσει στο δημόσιο τομέα Πρόκειται λοιπόν για μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να είναι μια μη αντιστρεπτή μεταρρύθμιση για την ε, διακυβέρνηση της χώρας μας. Δεν έχουμε βέβαια μόνο αυτά τα σχέδια για υποστήριξη του προϋπολογισμού, έχουμε μεγάλη υποστήριξη από ένα ειδικό εργαλείο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες από το τέλος του 2014 από ό,τι κατανοώ, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να έχει μια ειδική μονάδα για τα θέματα αυτά και έχουμε λοιπόν αυτούς τους ειδικούς εμπειρογνώμες που έχουν έρθει στα Υπουργεία μας και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές μας αιτήσει και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία που είναι εν εξελίξη. Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η διαδικασία υποστήριξης, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τα χρήματα που δίνονται στην κυβέρνηση, αλλά και από την ποιότητα των εμπειρογνωμόνων που έρχονται στη χώρα μας. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Συγχρόνως όμως, μπορεί να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα σε ένα τομέα και λιγότερα σε άλλους, αλλά δεν είναι το θέμα του, της υποστήριξης, αλλά του ρυθμού πρόοδου. Έχω ένα συνάδελφο εδώ, που είναι υφυπουργός για τα θέματα γεωργίας. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα χάρη στην βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης και των εμπειρογνωμόνων που μας έχουν βοηθήσει σε μια συνολική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα. Αυτό είναι μια διαδικασία της διαδικασίας ε, θέσης σε καθεστώς αγοράς όλων των προϊόντων μας, των αγροτικών προϊόντων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βοήθεια λοιπόν αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για κάθε τομέα και για κάθε κεφάλαιο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο λεπτομεριακές συζητήσεις για αυτά τα θέματα, αλλά γενικά εμείς χαιρόμαστε για τις απόψεις σας, για την εμπειρία που μεταλαμβαδεύετε και θέλουμε να τονίσουμε την μεγάλη συμβολή του Επιτρόπου Χάν και τη βοήθεια των υπουργικών των κλιμακίων που έρχονται από Υπουργεία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο εύκολο να συνεργαζόμαστε με αυτές τις χώρες, ιδίω από χώρες που αντιμετωπίσανε αντίστοιχα προβλήματα πριν από 5 πριν από 10 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά ήταν στην ίδια σελίδα με εμά και είχαν την ίδια διαδικασία αρρωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα εργαλεία τώρα τα οποία έχουν αναφερθεί, η ειδική μονάδα υποστήριξης στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο μας έχει παράσχει μεγάλη <clears throat> υποστήριξη σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση για τα θέματα της ε, δημόσιας διοίκησης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περισσότερη αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και, τον, και το κράτος δικαίου. Ήταν πολύ καλή συνεργασία μας με αυτό το ειδικό εργαλείο που έχει ανταποκριθεί στην υποστήριξη του γραφείου της εισαγγελία και ίσως οι αρμόδιοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορούν να προσθέσουν κάτι για το θέμα αυτό. Όπως είπε και ο κύριος Σάιρους Βόλσκι, ήταν μια σύσταση από το κοινοβούλιο μας πριν από ένα χρόνο να υπάρξει βελτίωση του μηχανισμού συντονισμού με το να δημιουργηθεί στην κυβέρνηση μια τέτοια μονάδα συντονισμού. Είναι δύσκολο να σας παρουσιάσω την αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου για το οποίο εγώ είμαι, ενός φορέα για τον οποίο εγώ είμαι αρμόδια. Αλλά σε ό,τι αφορά την ε, κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης, έχουμε μια καλύτερη μορφή συντονισμού, είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά στον Πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλα τα πολιτικά θέματα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να τύχει και αναδιάταξης για να έχει ένα ευρύτερο χαρακτήρα και καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εφαρμογής Λαμβάνοντα υπόψη το ρυθμό τη διαδικασία προσέγγιση και την εφαρμογή τη ατζέντα της Συμφωνία Σύνδεσης. Μέχρι στιγμή όμω αυτό ο φορέας έχει αναπληρωτέ υπουργού οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τα ευρωπαϊκά θέματα. Η προσέγγιση αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική, υπέρ δηλαδή των ευρωπαϊκών θεμάτων. Η καλή σχέση με τη δίκηση και τη δικιά μας αντιπροσωπείας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε, σε εργασιακό επίπεδο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε όλες τις συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Μεταρρυθμίσεων υπήρχαν εκπρόσωποι των ε, κύριων ε, κομμάτων του Κοινοβουλίου για να συζητηθεί η μεταρρυθμιστική ατζέντα. Μία φορά το μήνα λοιπόν, τουλάχιστον, εγώ συζητάω το θέμα της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Άρα υπάρχει συνεχής έλεγχος από όλε τις πλευρές, από τρεις πλευρές, και από το Κοινοβούλιο και από τον Πρόεδρο και από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ μας και με το Κοινοβούλιο και με τον Πρόεδρο για να τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία σύνδεση. Κάποια προβλήματα, όπως ακούσαμε, υπάρχουν στο Κοινοβούλιο, αλλά σε ένα βαθμό, το είπαμε και πολλές φορές σήμερα, το ακούσαμε, ότι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε είναι πολλές συγχρόνως και για τη δημοσιοδίκηση και για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Πράγμα που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο ετοιμάζει μια τεράστια ποσότητα νομοσχεδίων και νομοθετημάτων που είναι δηλαδή πάρα πολύ φορτωμένη. Γι' αυτό και υπάρχει μια δική διαδικασία συζήτησης κάθε νομοσχεδίου στη Βουλή μας. Είναι μια συνολική δουλειά που πρέπει να γίνει και από την κυβέρνηση και από το κοινοβούλιο, από κοινού. Αν μιλάμε για πακέτο νομοσχεδίων που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ή με άλλες συστάσεις για μεταρρυθμίσεις, πρέπει να ξέρετε ότι η συζήτηση γίνεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και η υπηρεσία που ασχολείται με αυτά τα θέματα έρχεται σε επαφή με τους βουλευτές για να συζητήσει τα νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία προσαρμογής Πολλές φορές επίσης αναφερθήκατε στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν κατά της διαφθοράς. Σίγουρα εδώ χρειάζεται μια τεράστια μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση αυτή κατά της διαφθοράς φυσικά πρέπει να αρχίσει και βήμα-βήμα να προχωρήσουμε σε δράσεις που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση αυτή. Γιατί όταν μιλάμε για την καταπολέμηση τη διαφορά, πρέπει να μιλήσουμε και για ιδιωτικοποίηση, πρέπει να μιλήσουμε για απορρίθμιση. Και εσεί πολλές φορές αναφερθήκατε σε μικρή πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές εξελίξεις επίσης επηρεάζουν την κατάσταση. Θα με διορθώσουν οι συνάδελφοι αν κάνω λάθος, αλλά το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης έχει Υπουργό υπεύθυνο για το κλίμα επενδύσεων, για την προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ήδη το Μάιο προτάθηκε μια τεράστια μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με την απορρίθμιση. Απλοποίηση δηλαδή ε, το πώ παίρνει άδεια μια επιχείρηση για να ξεκινήσει. Πιο απλέ διαδικασίε για τι επιχειρήσει, όχι μόνο τι Ουκρανικέ, αλλά οποιαδήποτε επιχείρηση που θα ήθελε να έρθει στην Ουκρανία. Αρχίσαμε λοιπόν αυτήν την διαδικασία και αναμένουμε απλοποίηση πάνω από 100 διαδικασιών. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα ή σε ένα μήνα, αλλά εφ' εξής, να ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε ε, την ε, τεχνολογία εχμής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για να επιφέρουμε αλλαγέ και στη λειτουργία του Υπουργείου Δικαιοσύνη. να μην υπάρχουν άμεσες επαφές με τον κόσμο που ζητάει άδεια, που ζητάει κάποια επίσημα έγγραφα από τους αξιωματούχου, αλλά να εφαρμόσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Και σε καθημερινή βάση, δύο-τρεις ώρες ασχολούμαστε με αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στην απορρίθμιση και τις οικονομικές αλλαγές. Μια στιγμή είναι εδώ που βρίσκομαι και να προσπαθήσω να συνεχίσω. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι εκείνη που έχει να κάνει με την αποκέντρωση και τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Για την αποκέντρωση. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που γνωρίζουμε. Τι έγινε στην Πολωνία, τι έγινε στη Γαλλία. Και ελπίζω να γνωρίζετε ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε συζήτηση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά με αλλαγές στο Σύνταγμα και την αποκέντρωση. Η αποκέντρωση είναι μια αποκέντρωση εξουσιών. Είναι μια διαδικασία που αρχίζει με την οικονομική αποκέντρωση. Άρχισε αυτό από την αρχή της χρονιάς, από 1η Ιανουαρίου του 2015. Ήδη μεταφέραμε κάποιες φορολογικές αρμοδιότητες σε τοπικές αρχές. Έξι μήνες τώρα. Μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι οι τοπικοί προπολογισμοί έχουν πάνω από 40% επιπλέον πόρους, αν τους συγκρίνουμε με το 2014, εξαιτία αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης και αποκέντρωσης. Έχουμε πρόβλημα με την οικονομική μεταρρύθμιση και τον οικονομικό τομέα, όπως αναφέρατε κι εσείς. Μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας, η κατάσταση στην Ουκρανία, Ανατολική Ουκρανία, μας κόστησε πάνω από το 20% του ΕΠ μας. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να σταθεροποιηθεί κάπως η οικονομική κατάσταση και το οικονομικό μας σύστημα. Μία από τις προτερότητές μας κατά της διαφθοράς στην ε, δημόσια δίκηση είναι η μεταρρύθμιση ακριβώς της δημόσιας δίκησης. Και θέλουμε να κάνουμε και μεταρρύθμιση στις τράπεζες για τη σταθεροποίηση της οικονομίας μας. Αν θέλετε οικονομικά δεδομένα μπορούμε να σας δώσουμε. Από τον Υπουργό Οικονομικών και Εμπορίου που είναι εδώ μαζί μου. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία του Μίνσκ. Εκτιμώ όλος ιδιαίτερο τη βοήθειά σας και τις κυρώσεις που επιβάλλατε κάθε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευπρόσδεκτη. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε, να θέσουμε σε εφαρμογή το δικό μας τμήμα, αυτό που αφορά εμάς στη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν είμαστε εμείς που σπάμε την συμφωνία, είναι η Ρωσία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν έρθουμε τώρα και αν ρωτάτε ποια είναι η, τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα για να βοηθήσει, το μόνο που μπορούμε να σας ζητήσουμε είναι να διατηρήσετε τις τρέχουσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές. Πολλές φορές ε, ρωτήσατε το θέμα διεθνών δράσεων υπό τον ΟΗΕ για να τεθεί σε εφαρμογή απόλυτα η συμφωνία του Μίνσκ. Οποιαδήποτε πολιτική και τεχνική στήριξη είναι ευπρόσδεκτη. Ξέρετε επίση ότι ως αποτέλεσμα των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και εδώ θέλουμε να στηριχτούμε στη δικιά σας βοήθεια για τους ανθρώπους που έχουν φύγει, έχουν μετατοπιστεί είναι πάνω από 1.300.000 από ό,τι υπολογίζουμε, που είναι κυρίως στο χάρτη και στο πετρόσκι. Και τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του πώς να βρουν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί, πώς ε, να τους αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που είναι εργατικό δυναμικό, το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, να υποφεληθούμε από αυτό στη χώρα. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν μένει ακόμα να το αντιμετωπίσουμε και ανθρωπιστικά αλλά και οικονομικά γιατί έχει και οι οικονομικές επιπτώσεις αλλά και κοινωνικές. Τώρα, τι είπατε για τον ιδιωτικό τομέα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να δώσω το λόγο στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό για τις εσωτερικές σχέσεις είναι εδώ στην ομάδα μας και μπορεί να σας απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ίσως καλύτερα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Όσον αφορά αυτήν την κατάσταση, είναι θέματα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα γίνονται έρευνες και ταυτόχρονα υπάρχει και μια διαδικασία διαμεσολάβησης. με άλλες δομές και με την ε, συμμετοχή όλων των αρχών επιβολής του νόμου. Αλλά είναι υπό την Ουκρανική κυριαρχία το όλο θέμα. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω το λόγο, να δώσω το λόγο και σε εκπροσώπους της Προεδρικής Διοίκησης. Για την ιδιωτικοποίηση επίσης νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει καλύτερα. Γεια σας να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε για όλα αυτά τα θέματα. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την συνεργασία επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης, Υπουργικού Συμβουλίου και Προεδρίας. Είναι επικοδομητική η συνεργασία που έχουμε και ενεργούμε σύντονοι και συμμορφούμε με το νέο σύνταγμα. Ενδεχομένως θα πρέπει να λιάνουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των παλαιότερων δομών και των νεωτέρων. Τώρα υπάρχουν καινούργιες αρμοδιότητε από πλευρά τη Προεδρία. Επίση υπάρχουν και κάποιε φήμε ε, για κάποια ολισθήματα τέλος των λάθος υπολογισμούς, αλλά δεν πρόκειται για κάτι το σοβαρό. Ε, προχωρεί η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε κάποιους νεοδιοριστέντες, οπότε και θεωρούμε ότι τώρα πρόκειται να συνεργαστούμε μόλις επιστρέψουμε στο Κίεβο. Θα συνεργαστούμε πιο αποδοτικά και θα φροντίσουμε τους ώστε να υπάρχει συνέργεια και όχι ανταγωνισμός μεταξύ κυβέρνησης και προεδρίας. Και φυσικά και Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, πρέπει να απαντήσουμε ένα άλλο ερώτημα. Πρόκειται για τη δεξιά. Δεν καταπολεμούμε κανένα φορέα, κανέναν πατριώτη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες προκλήσεις Και γίνεται αυτό από πλευράς των πολιτικών φίλων ή των πρώην φίλων. Τέλος πάντων. Υπάρχουν τώρα κάποιες παράνομες, κάποιες εγκληματικές δραστηριότητε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό αφορά κάποια συγκεκριμένα άτομα που ανήκουν στην δεξιά ή σε άλλους ε, φορείς, ακόμα και κάποιους που υπηρετούν στις διοικητικέ αρχές, στις τελωνιακές αρχές. Αυτό αφορά τα Καρπάθια και έχουμε ξεκινήσει ολόκληρη τη κατά πολύ της διαφθοράς. Οπότε. Και επίσης πρέπει να σας προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι ο αφοπλισμός της δεξιάς. Ο αφοπλισμός θα γίνει. Σύντομα, θα αφοπλιστούν από μόνοι τους. Μόλις αφοπλίσει η Ρωσία τους μισθοφόρους. Ευχαριστώ. Ο επόμενος. Ναι, αναφέρθηκε σήμερα ως μια πρόσθετη υπόθεση που έχει να κάνει με την ε, ιδιωτικοποίηση. Ήταν και μια αναφορά στην ομιλία του Πρόεδρου μας. Ήταν ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου ο οποίος τον προηγούμενο μήνα ανέπτυξε ένα πλήρες πρόγραμμα για την ε, ανάπτυξη στον τομέα αυτό, για την πρόθεση των επιχειρήσεων και του επιχειρήν. Δεν πρόκειται λοιπόν μοναχά για μια ανοιχτή ε, διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Δεν το βρίσκω αλλά για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της ε, ανοιχτής αυτής διαδικασίας με την συμμετοχή με διεθνείς φορείς οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία. Ίσως κάποιος συναδελφός μου από την Ουκρανική Αντιπροσωπεία θα μπορούσε να συμπληρώσει. Θα δώσω λόγο στον αρμόδιο Υπουργό Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ. Ίγκο Τόλγκοφ λέγομαι. Και χαίρομαι που είναι και πάλι. Να απαντήσω σε ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει τώρα άλλη ατζέντα για την κυβέρνηση της ε, Ουκρανίας από την ε, την ε, σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κύριο σημείο της δραστηριότητάς μας και στο Υπουργείο Άμυνας ασχολούμαστε συνέχεια με το θέμα αυτό. Κρυμαία επίσης είναι το επόμενο θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο Υπουργός Λαυρόφ της Ρωσίας είπε ποια είναι η θέση τους για την Κρυμαία. Αλλά για τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με τις κυρώσεις. Όσο εξακολουθεί η κατοχή της Κρυμαίας πρέπει να συνεχίσουν οι κυρώσεις γιατί η Κρυμαία είναι τμήμα του εδάφους της ε, Ουκρανίας για τις ρυθμίσεις της συμφωνίας του Μίνσκ. Αυτό είναι ένα σχέδιο του Πρόεδρου Ποροσέγκο, η βάση του σχέδιου Μίνσκ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο λοιπόν για μας. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο υποστηρίχθηκε από τους Ουκρανού, από το λαό τη Ουκρανία, γιατί κατέθεσε αυτό το σχέδιο για μια πολιτική και ειρηνική λύση. Δεν βλέπουμε άλλη λύση εκτός από πολιτική λύση. Για να φτάσουμε όμω στο κατάλληλο αποτέλεσμα χρειαζόμαστε και την απαραίτητη πολιτική θέληση στη Μόσχα. Δυστυχώ αυτό δεν ισχύει. Αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα είναι εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτα τα σύνορα ένα μεγάλο μέρος των συνόρων της Ουκρανίας στα Ανατολικά από τις Ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να μπαίνουν ε, ε, όπλα και χρήματα από τα σύνορα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μετακίνηση και αναδιάταξη των δυνάμεών τους, οι αποσχιστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε εχμαλώτους όπως προβλέπει η συμφωνία του Μίνσκ γιατί η ρωσική πλευρά δεν τηρεί τα υπεσχημένα. Να επανέλθω τώρα στο τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όπλα. Και τα ζητήσαμε. Όχι μόνο εδώ. Ζητήσαμε και σε διμερές επίπεδο και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει επίκαιρο χαρακτήρα Ίσως δεν λένε πολλοί ότι δεν είναι κατάλληλος, κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Αλλά η ρωσική πλευρά δίνει πυροβολικό και τάγκς στους αποσχιστές στην Ουκρανία κάθε μέρα. Δεν ρωτάνε κανένα το κάνω αυτό. Γιατί εμείς πρέπει να περιμένουμε. Τι πρέπει να περιμένουμε να συμβεί. Προτού δοθεί η απόφαση να υποστηριχθεί η Ουκρανία με όπλα και πυρομαχικά για να μπορέσει να υπερασπιστεί το έδαφος της. Μην ξεχνάτε ότι λοιπόν για μας αυτό είναι ένα κέριο θέμα. Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας. Και πάλι τονίζω ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ισχυρό στρατό ο οποίος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τι εισβολές. Έχουμε περίπου 60.000 μάχημα στα θέματα. Ξεκίνησαν πριν από 15 με 5 έως 7.000. Έχει γίνει λοιπόν τεράστια ε, βελτίωση χάρη και τη δική σας υποστήριξη. Και βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και στο μέλλον. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή με τη βοήθεια εκπαιδευτών από τον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Σουηδία, που θα έρθουν το Σεπτέμβριο για να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματα του, της Ουκρανίας επί τη βάση των προτύπων του ΝΑΤΟ. Επιλύουμε λοιπόν δύο προβλήματα έτσι, τη μεταρρύθμιση του τομέα άμυνας και την προσέγγιση του τομέα άμυνας και ασφάλειας Ουκρανίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα για την Ουκρανία είναι ότι πρέπει να επιτύχουμε την εδαφική μας ακαιρεότητα. Η Κρυμαία είναι υποκατοχή και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας βρίσκεται κάτω από επίθεση. Αν δεν λυθεί αυτό το θέμα δεν θα μπορέσει να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη και μην το ξεχάσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Νόμιζα ότι είχατε αναλάβει εσείς την προεδρία της συνεδρίασης. Υπάρχουν άλλα περαιτέρω θέματα. έχετε το λόγο. Η Αναμαρία. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχα τη δική μου έκθεση σε μια άλλη επιτροπή. Εγώ χαίρομαι που είναι παρόν. παρόντες οι αναπληρωτές υπουργοί. Πολλοί από εμά έχουν υποστηρίξει ιδιαίτερα την προσπάθεια του να γίνει κατανοητό ότι λαμβάνει η χώρα ένας πόλεμο στην Ευρώπη, υπάρχει πόλεμο επιθετικός παραβίαση του διεθνού δικαίου και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη υποστηρίζοντας τις κυρώσεις και τις συμφωνίες του Μίνσκ και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και το θέμα της Κρυμαίας. Προσπαθήσαμε επίσης να καταγγείλουμε την πάρα πολύ αρνητική ανθρωπιστική κατάσταση που ισχύει στην χώρα σας. Είχαμε επαφές με τον αρμόδιο επίτροπο του Χρήστο Στυλιανίδη όταν, όταν γύρισε από την Αποστολή Βοήθειας Έχουμε λοιπόν υποστηρίξει την βοήθεια από την ανθρωπιστική μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΕΚΟ και προσπαθούμε να αυξήσουμε και το προφίλ <clears throat> της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Βάσης στην Ουκρανία για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Θέλω να συγχαρώ την κυβέρνηση της Ουκρανίας και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας για την πάρα πολύ σημαντική τους δέσμευση σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή όταν υπάρχει πρόβλημα προσφύγων και πολέμου και όταν αντιμετωπίζει και την επίθεση και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου για το γεγονός ότι προχώρησε σε τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ιδίως για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει η υποστήριξη προς εσάς παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι τώρα διχασμένη. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και με την κυρία Μογκερίνη για να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση της προπαγάνδας με στοιχεία και με την αλήθεια. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ε, κάποια ερωτήματα τώρα τα οποία ίσως κάποιοι άλλοι τα έχουν θέσει. Το θέμα της εξάρτησης από ενεργειακούς πόρους και παροχή φυσικού αερίου ενώ πλησιάζει ο χειμώνα και επίσης και το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο τμήμα της ε, χώρας το οποίο δεν επηρεάζεται από την ένοπλη σύγκρουση, τι περαιτέρω θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Σύνδεσης και να αντιμετωπιστεί το κύμα προσφύγων το οποίο έχει ιστορικό χαρακτήρα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει λόγος να πρέπει να δευτερολογήσω ενώπιον σας, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που μόλις μετεδόθησαν, ο πρέσβης ε, Ελισέγεφ ορίστηκε ως μέλος της Προεδρικής Υπηρεσίας, οπότε θα πρέπει τον κύριο Ελισέγεφ να τον συγχαρούμε, γιατί είναι ο κατάλληλος και κατάλληλη θέση και θα είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας ε, μαζί του. Και θα έχουμε επίσης και κάποιον διπλωμάτη Ουκρανό που να είναι αποτελεσματικό, να μπορεί να επικοινωνήσει σωστά και πότε θα είναι ένας ε, εταίρος, ε, ένας συνεργάτης πολύτιμος εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό ήθελα πρόεδρε. Uh, Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα έναν καινούριο συνεργάτη, όπως αναφέρατε την κυρία Γκνίδιου, και Οπότε έτσι θεωρούμε θα είναι καλύτερη η συνεργασία με τον κύριο Ελισέγιος, γιατί έχει τεραστία εμπειρία. Ξέρει από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και ελπίζουμε η πως να πιάσει τόπο στην Ουκρανία όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Όσον αφορά την ερώτησή σα, γιατί έχουμε του συναδέλφου που ασχολούνται με κοινωνική πολιτική που είναι εδώ και εσεί είπατε το πρόβλημα αυτό για αυτούς τους 3.000 που χρήζουν βοηθείας. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτά τα οριστικά αριθμητικά στοιχεία. Γιατί έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από το Λουχάνσκ και το Ντονιέσκ. Αυτοί έχουν καταγραφεί, υπάρχουν στο σύστημα, αλλά η επιβίωσή τους γίνεται μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας. Επίσης, το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο προτείνει για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τους εκτοπισμένους. Και πάρα πολλοί εκτοπισμένοι βρίσκονται ακόμα στα κατεχόμενα. Και τώρα δίνουν τη σκητάλη στον αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την κοινωνική πτυχή τους. Έχετε το λόγο. είναι ο Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων. Ενάμιση λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Και μετά η κυρία Ρούτιτσκα. Παρακαλώ. Είναι ο κύριος Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ξέρετε όμως, τα θέματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα για την Ουκρανία στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Όμως, για τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της χώρας μου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι πρέπει να ευθώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα εργασιακά και άλλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση στην Ανατολική ε, Ουκρανία μας ε, οδηγεί σε επιπλέον δυσκολίες εργασιακά, γιατί όπως είπαμε είναι πάνω από ένα εκατομμύριο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, φύγει από τις περιοχές τους και για αυτούς πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προστατεύσουμε κοινωνικά. Οι εσωτερικά λοιπόν μετατοπισμένοι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και 3,4 δις έχουμε δώσει ουκρανικές κόνες για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα των μετατοπισμένων, γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να περάσει προγράμματα για την προστασία τους και για την ένταξή τους τις επόμενες χρονιές. 2015-2016 είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί στα κυβερνητικά σώματα. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, το κύριο μήνυμά μου για να απαντήσω τι περιμένουμε από την ευρωπαϊκή πλευρά, η απάντηση είναι ότι μετά την κατάσταση αυτή που έχουμε με τους εκτοπισμένους εσωτερικά, έχουμε πρόβλημα με τις εργασιακές ρυθμίσεις και πρέπει να υπάρξουν μέτρα για να προωθήσουμε την απασχόληση του πληθυσμού αυτού. προσπαθούμε να εισάγουμε προστατευτικούς μηχανισμούς για αυτούς τους ανθρώπους και η ανθρωπιστική αρρωγή φυσικά και χρειάζεται. Επιπλέον όμως αυτό που ζητάμε είναι σχεδιασμό προγραμμάτων ώστε να υπάρξει περισσότερη αποσχόληση για τους ανθρώπους αυτούς στην Ουκρανία γιατί είναι ήδη μαζεμένοι σε κάποιους οικισμούς, επιπλέον όμως πρέπει να υπάρξει απασχόληση για να ενταχθούν στην Ουκρανική κοινωνία. Αυτά, εφόσον δεν έχουμε χρόνο, σταματάω εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, εσείς τώρα. Ευχαριστώ. Είμαι αναπληρωτής ε, υπουργό για τα θέματα ευρωπαϊκών ζητημάτων που έχουν να κάνουν και με τη διατροφή. Έχουμε συνεργαστεί πολύ μεταξύ μας μέχρι τώρα για την εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται στην Συμφωνία Σύνδεσης. Είμαστε ένα βασικό Υπουργείο για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Και γι' αυτό, αυτό που θέλουμε να σας ζητήσουμε, όταν ρωτάτε τι βοήθεια χρειαζόμαστε, ε, λοιπόν χρειαζόμαστε στήριξη για την ε, επικαιροποίηση της νομοθεσίας μας, ώστε να πάει στο Κοινοβούλιο και να περάσει. Το τελευταίο εξάμεινο δουλέψαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια συνολική στρατηγική όσον αφορά την γεωργία. Τώρα σε εθνικό επίπεδο θα πάει τι διοικητικές υπηρεσίες της Προεδρίας για να προχωρήσει η αναθεώρηση, να πάει δηλαδή και στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Μετά θα περάσουμε στην εφαρμογή. Οπότε, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική. Κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου μας, ε, Γεωργίας και Τροφίμων, είναι να υπάρξει κτηματολόγιο για την αγροτική γη. Ευχαριστώ. Τα τελευταία, τελευταία, τα τελευταία λόγια τώρα. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση στην ε, ρωσική επίθεση είναι οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε στη χώρα μας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λίγη συνεδρίαση. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να συναντηθώ με την Επιτροπή Περιπολογισμών, γιατί αν δεν υπάρχει δικιά του στήριξη, ξεχάστε όλα αυτά που μας ζητάτε. Δεύτερον, προτείνω την επόμενη φορά να συναντηθούμε με τους αναπληρωτές υπουργούς. Μαθαίνουμε περισσότερα από ό,τι με τους ίδιους τους υπουργούς. Αυτή είναι η εντυπωσή μου από τη σημερινή συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Μπάλας για τη συμμετοχή σας. Καλή όρεξη.